We believe that we can start because we are a little bit delayed. Καθυστερήσαμε λίγο, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε ε, την ακρόαση για τα drones, τα μη πανδρομένα αεροσκάφη. Yeah. Όσοι, όσοι πρέπει να παρίστανται. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα της διάταξη είναι να ναι, ζήτησα από τους συνεργάτες μας να μου πούν να αρχίσουμε. Αγαπητοί νεαροί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα μας είναι η έκθεση της κυρίας Γκόμες σε δεύτερη ανάγνωση για τη θαλάσσια διάσταση της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Ελπίζουμε ότι και οι σκιώδεις ηγητές ήταν εδώ. Οι Γκόμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συμβολή τους σε αυτή την έκθεση, για τις ε, τόσο ουσιώδεις ε, τροπολογίες που έχουν υποβάλει. Δεν τις έχω δει όλες, αλλά επεξεργάστηκα 19 συμβαστικές τροπολογίες μόνο. Και χθες τις ε, διαβίβασα, οπότε οι δεν θα έχουν προφτάσει να τις διαβάσουν, αλλά από ό,τι ξέρω θα τα πούμε στο Στασβούργο, τόσο ώστε να συζητήσουμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ είμαι ανοιχτή. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ επικοδομητικές αυτές οι τροπολογίες σε γενικές γραμμές συμφωνούμε, οπότε και προσπάθησα να συμπεριλάβω όλες τις τροπολογίες στις συμβαστικές διατάξεις, γιατί θεωρώ ότι αναβαθμίζουν, βελτιώνουν την έκθεσή μου. Σε κάποια σημεία δυσκολεύτηκα λίγο περισσότερο. Έχουμε και τις προτάσεις του κυρίου Μπουτικόφερ. Θα, όσο μπορώ, όπω είπε ο κύριος Μπουτικόφερ, θα τα περιλάβω. Πάντως, σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τον κύριο Ντόν τη Λίζα, διότι δουλέψατε σκληρά και οι τροπολογίες είναι πολύ ουσιαστικές. Και εγώ η ίδια συνέταξα κάποιες τροπολογίες επί τη βάση των όσων αξιόλογων είπαν διάφορες ε, υπηρεσίες και έτσι βελτιώνω το αρχικό μου κείμενο. για τα υπηρεσίε, ενώ ας πούμε την, Ευρω... την υπηρεσία εξωτερική δράση, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα κλπ. Τώρα υπάρχει ένα τομέα όπου θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο Στασβούργο. Τι θα πούμε και πώς θα το διατυπώσουμε για την Αρκτική. Ναι, δεν υπάρχουν τίποτα άλλα προβλήματα. Και θεωρώ ότι θα συγκεντρώσουμε τη Γενική Συνένεση. Και έτσι θα βάλουμε το λιθαράκι μας στην προετοιμασία της Υπουργικής Συνόδου ε, για τη θάλασσα και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Θάλασσας του Δεκεμβρίου. Άνα σε ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Κύριε Λίζα, γιατί τώρα λόγο και αντικαταστάτε τον κύριο Ντονζό. Ναι, για δύσκολο γιατί έχει κάποια άλλη υποχρέωση ο κύριο Ντονζό, δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε μου ζήτησε να διαβάσω τι δικέ του παρατηρήσει και θα το κάνω μεγάλη μου χαρά πρώτα-πρώτα. Εκ μέρου του κύριου Ντονζό, συγχαρητήρια κύριε Αγκόμε για την έκθεσή σα. Μα ε, δίνετε μια πλήρη εικόνα των κινδύνων, των απειλών, τη ε, ασφάλεια από πλευρά θάλασσα και να δούμε επομένω τι στρατηγική θα μετέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού του κινδύνου και τι απειλέ. Και ο κύριο Λεωνζό είπε και στην πρώτη συζήτηση που έγινε για την έκθεση κυρία Γκόμε, το μήνυμα λέγει θα μπορούσε να είναι πιο δυναμικό ε, και πιο σαφέ και αυτό μπορεί να γίνει με κάποιε τροπολογίε. Υπέβαλε 47 τροπολογίε στο κείμενό σα. Τώρα ποιο είναι ο σκοπό των τροπολογιών. Πρώτον, να αλλάξει η εστίαση ε, τη έκθεση. όπως εξήγησε στην τελευταία μας συνάντηση του κ. Ντανζόν παρά το ότι ο τίτλο τη έκθεσης είναι η θαλάσσια διάσταση της ΚΕΠΑ η έκθεση επικεντρώθηκε περισσότερο στον ορισμό μιας ευρωπαϊκής θαλασσίας στρατηγικής. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα μέσα της ΚΕΠΑ σε σχέση με την ΚΕΠΑ την ίδια, γιατί θα πρέπει να θεωρήσουμε το ότι θα πρέπει να εξελιχθούν και αυτά τα μέσα πολιτικές και έτσι να εξασφαλίσουμε την ε, θαλάσσια ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε μια σειρά τροπολογιών επομένω, ούτω ώστε προσπαθούμε να προστεύσουμε την έκθεση και ε, σύμφωνα με τον κύριο Ντονζόν η έκθεση πάσχει γιατί είναι πάρα πολύ λεπτομερής και πάρα πολύ μακροσκελής. Έχουμε εδώ επίσης μια σειρά άλλαγων στην σειρά των να κείμενο και έτσι να έχουμε μια επιχειρηματολογία πιο ξεκάθαρη. Επίσης, σε διάφορες από αυτές τις τροπολογίες ε, προσπαθούν να αποφύγουν τις περίτες επαναλήψεις, γιατί πολλές παρέφυλα το ίδιο πράγμα. Έχουμε επίσης πάρα πολλές τροπολογίες για διευκρίνηση των λέει το κείμενο και ε, ο κ. Ντομζό επίσης προσπαθεί να σταθεί ε, τι γίνεται όσον αφορά τη, την, τη, τη του συστήματος, επίσης και την ασφάλεια μπορεί να, να παράσχει το, το κράτος. Έχουμε επίσης, σε σχέση με αυτό την τροπολογία 20, ε, όσον αφορά τη στρατηγική της Θάλασσα για την Ευρώπη, εδώ ο κ. Ντονζόν θέλει να ξεκαθαριστεί ποια μέτρα στατικής μπορούμε να μετέλθουμε και επίσης έχουμε σχετικά εδώ την τροπολογία 57 Τώρα, ε, εδώ στις ε, ε, απειλές, αναφέρει και στον Ζώο, ποιες θεωρείται είναι αυτές οι απειλές, οι συμβατικές, τροπολογία 66, επίσης σε κάποιο τρομοκρατικού χαρακτήρα απειλές, στο 74 πειρατεία, το 80 και επίσης η ΚΕΠΑ, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές στην τροπολογία 81. Τώρα, έχουμε κάποιες άλλες ε, τροπολογίες και εξηγεί ότι ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός είναι χώροι θαλάσσιας αστάθειας. 106, 107 και 127 είναι σχετικές τροπολογίες. Επίσης, εκφράζει την απειλή ότι θα πρέπει να έχουμε εταιρικές σχέσεις με κάποιες με κάποιες, συνεργασίε με κάποιε χώρε τρίτε, όπω λέει στην Τροπολογία 125, όπω είπε η κυρία Γκόμε, χθε το απόγευμα ε, λάβαμε τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε και τι μελετά σε συνεργασία με το επιτελείο σα και εσά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνεργασία σχετικά με τα περισσότερα από αυτά. Ευχαριστώ. Άννα, σε συγχαίρω εκ μέρου τη για την έκθεση αυτή. Ε, είναι πολύ καλή, ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη, εντάξει, πολύ καλή. Αντιμετωπίζεις όλα τα ζητήματα. Αυτά που συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συζητηθούν σε μια τέτοια έκθεση. Έχω μερικά πράγματα να πω μόνο. Χρειάζεται θαλάσσια στατικική. Πολύ καλά το αναφέρει. Είναι πλήρης η προσέγγιση. Καλύπτει κάθε απειλή και πρόκληση. Καλό αυτό είναι μια πολυτομιακή προσέγγιση. Χρειάζεται αυτή η προσέγγιση όταν μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια και μια σχετική έκθεση. Αναφέρθηκε στους κινδύνους και την τρομοκρατία, τις εγκληματικές πράξεις, αναφέρθηκε στις διάφορες περιοχές που έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν κινδύνους όπως η θάλασσα της Κίνας, η νότια θάλασσα της Κίνας ε, και έχουμε υποβάλει τροπολογίες σχετικές. Ευχαριστώ που δέχθηκες τις τροπολογίες που αφορούν τον εύξηνο πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα. Ε, οι Ρουμάνοι και κάποιος από τη Βουλγαρία συνάδελφος ασχολήθηκε με το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι ο εύξηνος πόντος είναι πράγματι πολύ σημαντικό θέμα από πλευράς ε, ασφαλείας. Κοιτάξτε τι, έχει, τι συμβαίνει. Και επίσης ομαδοποίηση των πόρων, μοίρασμα των καθηκόντων, το pooling and sharing, ε, συνεχίζει την προσέγγιση μας για την ΚΕΠΑ. Πολύ καλό αυτό. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά τις συμβαστικές λύσεις και θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ καλή έκθεση και πραγματικά αναγκαία. Μέχρι τώρα δεν αναφερόμαστε εκτενώς στη θαλάσσια διάσταση, αλλά στο μέλλον, το μέλλον του κόσμου είναι στη θάλασσα και στο διάστημα. Ο κύριος Βαν έχει διαφορετική άποψη και θα πάρει και το λόγο. Um, Όπως βλέπετε, ο Ράιναρντ Μπίτιχόφερ έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες και οι πράσινοι πιθανότατα κρύβονται πίσω από αυτές. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, είναι πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα το κείμενο. Είναι πολύ καλό, σαν να είναι από καλό συγγραφέα. Και βλέπουμε ότι εμφανίζονται και περιοχές του κόσμου και τονίζονται στην έκθεση. Είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση αυτή και τις τροπολογίες Πέτι Χόφερ. Ο κ. Βανόρντεν. Η Βρετανική προσέγγιση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κανείς δεν υποτιμά τη σημασία των θαλασσών και της ελεύθερης ναυσιπλοίας και των εμπορικών ε, δρόμων. 75% του εμπορίου μετακινείται θαλασσίας οδού. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες μας. Είναι ζωτική σημασία. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό. Το θέμα είναι ε, ποια είναι η θαλάσσια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, βέβαια είναι, αφορά την ΚΕΠΑ ουσιαστικά. Προσθέτουμε, στολίζουμε την ε, ήδη υπάρχουσα τεκμηρίωση για την ΚΕΠΑ. Αν θεωρούσα ότι θα παραχθεί άλλο ένα πολεμικό σκάφος λόγω της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, θα είχα διαφορετική άποψη. Όμως, τίποτα παραπάνω δεν παράγεται. Δεν υπάρχει η παραμικρή προστιθέμενη αξία από την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ενώσης από τα ζητήματα. Χαίρομαι που θεώρησε η Άννα ότι οι τροπολογίες μας ήταν επικοδομητικές. Και εγώ θεωρώ ότι οι δικές μου είναι επικοδομητικές, αλλά αμφιβάλλω ότι θα τις δεχτεί όλες. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να αφαιρέσω αναφορές σε υπερβολικές και άσχετες φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τόνισα τον ΝΑΤΟ, έθεσα την προσοχή, την προσοχή για τον ΝΑΤΟ, αλλά συγχαίρω την Άννα για ένα σημείο που αναφέρει για την 117. Την προτείνω, την υποστηρίζω την 117. Μιλάει για την καταπολέμηση της πειρατείας. Η πλέον επιτυχής, ο πλέον επιτυχής παράγων για, το, για να δαμαστεί το φαινόμενο της πειρατείας δεν ήταν η εμπλοκή ε, ναυτικών πολεμικών σκαφών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά η χρήση ιδιωτικών φυλάγων, ιδιωτικών αρμοδίων για την ασφάλεια από ιδιωτικές εταιρείε. Και αυτό είναι ο σημαντικότερος ιδιωτικός παράγων για τη μείωση της πειρατείας. Και η τροπολογία μου συγκεκριμένα το παρουσιάζει, το εισάγει αυτό. Ελπίζω να το λάβει υπόψη, Άννα. Είναι η τροπολογία μου 117. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Λούζινγκ. Ήδη τα είχα πει όλα την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό να δώσετε τώρα το λόγο στον κύριο Αγκουράκη. Ah. Κύριε Αγκουράκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εμείς ε, είμαστε αντίθετοι με την έκθεση. Δεν θα μπω σε αυτά και είμαστε αντίθετοι γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικό βήμα στην στρατιωτικοποίηση γενικά των διεθνών σχέσεων και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα αστάθειας, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Ε, για μας η ουσία της έκθεσης βρίσκεται σε αυτό που σημειώνεται σε κάποιο σημείο στην αρχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε αισθάνονται ότι περιορίζεται η πρόσβασή τους σε παραδοσιακές θαλάσσιες περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πάνω σε αυτό το πράγμα τώρα οικοδομείται μια ολόκληρη ιστορία. Που βέβαια είναι ένα θέμα. Τι στο διεθνείς σχέσεις θα κάνουμε και πόσο ισότιμες θα είναι αυτές εάν η θαλάσσια πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να προστατεύσει τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους μόνον ενάντια στους ανερχόμενους Ρώσους, Κινέζους, Βραζιλιάνους και Ινδούς ενδεχομένω, δεν ξέρω άλλοι. Και για να δείτε όμως πόσο δύσκολα και επικίνδυνα είναι τα πράγματα, θα αναφερθώ μόνο σε δύο από τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, ε, γιατί τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Καταρχήν, ξανά υπάρχει ένα θέμα στην τροπολογία ε, συμβαστική, την τροπολογία 3, ε, επανέρχεται το θέμα των απειλών να, με, να μου επιτρέψει κυρία Γκόμες να διαφωνήσω με το θέμα των απειλών <laughs> διότι οι απειλές που έχουν σχέση με τη φτώχεια και με μειωμένο κρατικό έλεγχο και με μειωμένες δυνατότητες ε, επιβολής του νόμου δεν είναι καινούργιε. Αυτές είναι πάρα πολύ παλιές. Δεν είναι κάτι το καινούργιο που υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι και η έκθεση όμως δεν παίρνει θέση και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει ένα θέμα, είναι αυτό που λέει ότι είναι κατακαιρματισμένος ο θαλάσσιος έλεγχος σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όντως. Αλλά αυτό δεν μας το εξηγεί η έκθεση παρακάτω. Πού είναι ο κατακαιρματισμός, γιατί είναι κατακαιρματισμός, τι μέτρα θα πάρουμε για τον κατακαιρματισμό. Επειδή ακούστηκε κάτι για την πειρατεία, εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω εάν μειώθηκε ή δεν μειώθηκε λόγω της παρουσίας ε, ιδιωτικών ομάδων ασφαλείας στα πλοία. Αυτό όμως που ξέρω εγώ είναι μπορεί να μειώθηκε κάπως στη Σομαλία, αλλά μας βγήκε στην Δυτική Αφρική η πειρατεία και μπορεί να την μειώσουμε και εκεί θα μας βγήκε κάπου αλλού. Ε, τι θα γίνει, θα κυνηγάμε αυτό παντού. Και για να μην σας κουράσω ακόμα περισσότερο, θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο και θα σας το πω ευθέως, απαράδεκτη μία διατύπωση που μπήκε στην ε, τροπολογία 3, η οποία λέει ότι η σημερινή κατάσταση κάνει όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίζουμε ποιες είναι οι νόμιμες από τις παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε τι λέμε με αυτό το κείμενο. Στην αρχική, στο αρχικό κείμενο της κυρίας Γκόμες υπήρχε κάτι πιο σωστό και πιο σοβαρό, εν πάση περιπτώσει. Έλεγε ότι αυξάνουν και οι νόμιμες και οι παράνομες. Και εντάξει, να δούμε ποιες είναι οι παράνομες. Αυτό που λέει τώρα η τροπολογία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίζουμε τις νόμιμες από τις παράνομες, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι αυτός που έχει τη δύναμη θα θεωρεί ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο και τελείω η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, η κυρία Τζαβέλα. το Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Άννα, όπως πάντα η έκθεση της και το κείμενό της είναι πολύ καλό. Ε, αν είναι μακροσκελές, πιστεύω ότι είναι το θέμα τόσο σημαντικό και θα έπρεπε πράγματι να αναφερθεί σε πολλά θέματα. Ε, το πρώτο σημείο που θα θέλαμε να ε, επισημάνουμε είναι ότι πράγματι μας λείπει μια, ευρωπαϊκή, ε, μια πολιτική ευρωπαϊκής θαλάσσιας ασφάλειας. Ο κατακαιρματισμένος θαλάσσιος έλεγχος προκαλεί και είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Αραβική Άνοιξη στην ε, Βόρειο Αφρική έχει φέρει πολλές αλλαγές στη Μεσόγειο Είπε ο κύριος Αγκουράκη ότι η έκθεση ζητά μια στρατικοποίηση των διεθνών σχέσεων. Ο πλανήτη μας δυστυχώ υφίσταται κάθε είδους απειλές. Οι απειλές αυτές μπορεί να είναι και φυσικές καταστροφές. Μπορεί να είναι απειλές ε, κατά της ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρο μέρος των κρατών μελών ε, είναι βρέχεται από τη θάλασσα. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία πράγματι ζητούν μία κάλυψη ευρωπαϊκή. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία επιχειρούν να αξιοποιήσουν τον ενδογενή πλούτο που βρίσκεται στη θάλασσα, που μπορεί αυτός να είναι η αλία, και τα οποία ζητούν την προστατευτική ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της πειρατείας είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέλθει είτε όπως το βλέπουμε στη Σομαλία αλλά και να είναι επακόλουθο εσωτερικών εθνικών ε, διαμαχών όπως στη Λιβύη. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό ότι η Λιβύη αυτή τη στιγμή έχει έναν σχεδόν εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχει πειρατικό στόλος της Λιβύης, ανοιχτά της Λιβύης, ο οποίος απαγορεύει την ανθρωπιστική βοήθεια να πάει στη Βεγγάζη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη θαλάσσια ασφάλεια και επίσης να καθορίσει τα μέσα και τους τρόπους και τη στρατηγική η οποία θα αφορά αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική για τη θαλάσσια ασφάλεια. Στο, στην παράγραφο 3 συμφωνούμε με αυτό που είπε ο κύριος Αγκουράκης. Ήταν πολύ πιο σωστό το αρχικό κείμενο της κυρίας Γκόμες από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στην ε, τροπολογία. Και επίσης θα έλεγα ότι στην τροπολογία 14 έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι η καλύτερη ε, διατύπωση γιατί αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση αυτή τη στιγμή σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Fragmented. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα σχόλια. Όπως είπα, θα ήθελα το κείμενο να είναι όσο συνενετικό, όσο περισσότερο συνενετικό γίνεται, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να δώσει πραγματικά ένα μήνυμα και να επηρεάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική ναυτικής ασφάλειας. Σχετικά τώρα με τα σχόλια που άκουσα, Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένα, ορισμένες από τις τροπολογίες που έχει πάλι ο κ. Ντανζάν και άλλοι στοχεύουν στο να αφαιρέσουν ορισμένα ίσως λιγότερο χρήσιμα πράγματα από το κείμενο και εγώ κάνω μια προσπάθεια να το κάνω πιο λιτό και ευχαριστώ για την συμβολή σας. για τα όσα ε, δήλωσε ο κύριος Βαν Δεν συμφωνώ με την άποψή του για την μείωση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα, όχι τόσο να μειωθεί το νόημα της ε, ΚΕΠΑ, γιατί έχουμε και υπερεθνικές απειλές και γνωρίζω ότι αντιλαμβάνεται την ε, σημασία της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, αλλά ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουμε υπερεθνικές απειλές, καμιά χώρα από μόνη της δεν μπορεί αυτή να αντιμετωπίσει, ούτε το ίδιο το ΝΑΤΟ, παρόλο που αναγνωρίζω την ε, ε, δουλειά που κάνει το ΝΑΤΟ και έχω κάνει και αναφορές στο ΝΑΤΟ μέσα στο κείμενό μου, αλλά και το ΝΑΤΟ ακόμη μόνο του δεν είναι σε θέση να ε, χρησιμοποιήσει τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι απειλές αυτές. Γιατί δεν είναι και καθαρά θαλάσσιες οι απειλές και χρειάζεται και άλλη προσέγγιση. Και μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μπορεί να δράσει. Αυτό δε είναι το όραμα εντό εισαγωγικών προσπαθώ να προωθήσω με την έκθεσή μου. Και νομίζω ότι υπάρχουν και, υπάρχει και μεγάλη συμφωνία και από τις ε, τροπολογίες, το βλέπω αυτό που έχουν καταθέσει άλλες ε, πολιτικές ομάδες και ο κ. Νικολάη και το Λαϊκό Κόμμα και οι Πράσινοι. Η 117 στην οποία αναφερθήκατε είναι ωστόσο αρκετά περίπλοκη Εγώ δεν συμφωνώ με την ε, υποστήριξη της χρήσης ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας. Αλλά θεωρώ ότι γίνεται προσφυγή σε αυτές διότι δεν υπάρχει, διότι λείπει η παρέμβαση της κοινή εξωτερικής πολιτικής, της κοινής μάλλον πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Γι' αυτό καταλήγουν να βάζουν ιδιωτικού φρουρούς στα πλοία. Δέχομαι ωστόσο ότι αυτό συμβαίνει. Θα προσπαθήσω με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση συνδιαλλαγής να δεχθώ ότι αυτό συμβαίνει. Ό,τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτό αποτελεί ακριβώς απόδειξη του ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας που θα καθιστούσε την προσφυγή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας με όλα τα προβλήματα, όλη αυτή την πηξίδα της Πανδώρας που ανοίγει, θα την καθιστούσε απαραίτητη. Τώρα, για τα όσα δήλωσε ο κύριος Αγκουράκης. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν οι απειλές και ότι αυτές είναι και υπερεθνικές. Δυστυχώς γυρνάει πολύ μακριά από το μικρόφωνο, δεν την ακούμε καλά. Ο στόχος είναι να βασιστεί Δυστυχώ δεν την ακούμε καλά, δεν μπορούμε να σα μεταφράσουμε απολύτω αυτό που λέει. Είναι στραμμένη πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ, αύριο. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι όντω υφίστανται οι απειλές αυτές και ότι η απάντηση στις απειλές είναι κατακαιρματισμένη, είναι ασυνεχής, συχνά αντιφατική και ακόμα περισσότερα, περισσότερο συχνά αφήνεται στα χέρια διαφόρων χωρών μελών και μάλιστα αυτές δρούν με τρόπο που είναι ασύμβατος με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο λόγος που θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή η νέα προσέγγιση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι να βασιστούν αυτές οι απαντήσεις στις κοινέ αυτές απειλές όχι μόνο σε ένα λειτουργούν ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, με τις αρχές και τις αξίες του. Εγώ πιστεύω επίσης Βλέπετε και στου ίδιου μίλησατε για πειρατεία. Η δράση, η αντίδραση δηλαδή της Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών εταίρων υπήρξε επιτυχής. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτό το είδος εγκληματικότητα να πηγαίνει αλλού, σε άλλα μέρη του κόσμου. Και όχι στου ωκεανού που είναι τόσο σημαντικοί για την ελευθερία ναυσιπλοείας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό εργαλείο και προσέγγιση και μάλιστα που να αποτρέψει, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι συμφωνείτε, την προσφυγή, όπως βλέπουμε τώρα, έξω από τις αυτές της Ομαλίας, σε σκάφη εξοπλισμένα από και με ιδιωτικούς ρούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας που δρούν έξω από κάθε κανονιστικό πλαίσιο. Ακριβώς για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας. Τα προβλήματα δεν θα εξαφανιστούν, χειροτερεύουν. Και βλέπουμε ότι έφυγαν από τον Ινδικό ωκεανό και έρχονται κοντύτερα σε μας, στον κόλπο της Γουινέας. η διάκριση μεταξύ νομίμων και παρανόμων δραστηριοτήτων. Θα το κοιτάξω αυτό που είπατε και το είπε και άλλος ε, συνάδελφος. Ίσως χρειάζεται να διατυπώσουμε καλύτερα, να βελτιώσουμε τη διατύπωση εκεί. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τι εννοεί. Δηλαδή βλέπουμε όλο και περισσότερο να εμφανίζονται καταστάσεις όπου δήθεν νόμιμες δραστηριότητες στην ουσία είναι κάλυμα για παράνομες δραστηριότητες. δραστηριότητες. Πριν από λίγα χρόνια, για παράδειγμα, τα υποβρύχια ήταν καθαρά χρήση κρατική, έτσι, από κράτη, υποτίθεται σε νόμιμη δραστηριότητα. Βλέπουμε τώρα ε, συγγνώμη, υποβρύχια να τα χρησιμοποιούν λαθρέμποροι ναρκωτικών από τη Δυτική Αφρική και παίρνουν πορεία προς την Ευρώπη. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η διάκριση. Άλλο παράδειγμα, πρόσφατα ο αρχηγός του επιτελείου της Γουινέας Βισάου συνελήφθη από τους Αμερικανούς σε μια επιχείρηση σε διεθνή υδατά κοντά στη Γουινέα Μπισάου διότι συμμετείχε σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και είχε και σχέση και με την ΦΑΡΚ. Μα θα πείτε, ο επιτελάρχης του στρατού μιας χώρας, τέλος πάντων είναι μια αρχή ο άνθρωπος, είναι θεσμική, θεσμικό όργανο. Δυστυχώς, αυτή η χώρα τώρα πάει να γίνει χώρα λαθρεμπορίων ναρκωτικών με συμμετοχή των ανώτερων αρχών της χώρας αυτής σε λαθεμπόρια ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει η διάκριση αυτή. Και κάνοντας τη διάκριση αυτή βέβαια δεν θα μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε από την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου και άλλες βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι το σημαντική ως βάση. Γιατί αλλιώς κάποιοι θα κάνουν ό,τι θέλουν, κάποιες χώρες μέλη θα κάνουν ό,τι θέλουν, αναλόγως του αν θα είναι αυτά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή όχι. Παρατήρηση Βανόντων, χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Αλλά με την Ένωση πολλά έχουν επιτευχθεί και η ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άλλοι αλλού στρέφουν τα βλέμματά τους προς εμάς σαν πρότυπο. Εγώ συμμετείχα σε αντιπροσωπεία της οποίας ε, ηγήθη ο κύριος Μπροκ στη Βραζιλία όπου συζητήσαμε διεξοδικά με την, ε, με την βραζιλιάνικη κυβέρνηση και ένας από τους τομείς που τους ενδιέφεραν πάρα πολύ είναι τι κάνουμε εμείς στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, διότι τους απασχολεί. Και επειδή βρέχονται από τον Ατλαντικό, θεωρούν ότι έχουν ρόλο να παίξουν, επομένως και η ιδέα των συνεργασιών που τόνισαν και άλλοι από εσάς τις σας, είναι πολύ σημαντική για την Ένωση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει εκτός πλαισίου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και, δικαίου, και ιδίως του δικαίου της θάλασσας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς και η προσπάθειά μου αυτή θα είναι. Βέβαια, έχω τις απόψεις μου. Αλλά νομίζω ότι ευτυχώς συμπίπτουν με τις αντιλήψεις των περισσότερων μελών της Εποπιτροπής. Να, επομένως που είναι πάρα πολύ συναρπαστική η συζήτηση και αυτό αποδεικνύει πόσο, πόσο, πόσο ενδιαφέρον είναι να υπάρχει ποικιλία απόψεων. Οπότε είπαμε ότι με την ΚΕΠΑ έτσι γίνεται. Και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η πτυχία άλλωστε. Βέβαια, πρέπει κανείς να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι προβλέπετε, θα ψηφιστεί στις 35 η έκθεση 30 Μαΐου. Και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα... Καλώς ήρθατε ο φίλος. Μου επιτρέπετε να, το, ε, να σας αποκαλώ έτσι, μια που τόσο συχνά τα λέμε. E Είναι ο κύριος Παπόφσκι, ο νεκροτής γενικός γραμματέας τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Είχατε παραστεί στο Συμβούλιο των Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο στι 23 ε, Απριλίου. Oh, our uh, colleague is the Deputy Secretary General, but all of us we know uh, this. And we give... Και θα σας δώσουμε θέση αμέσω το λόγο. Thank you very much, uh, Madam, Madam Chair. Try again. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Υπουργή Αμήνης Δευτέρα και Τρίτη συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο σαν Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και υπήρξε δείπνο εργασία, κυρίως συζήτησαν για την κατάσταση στο Μαλί και είχαμε εισηγήσει του κυρίου Λεκουάντα που είναι επικεφαλής της Εκεί Δύναμης Επέμβασης Οπότε η αποστολή συνεχίζει να εξελίσσεται. Σύμφωνα με την εντολή, εκεί εκτελεί και εκπαιδευτικές δραστηριότητε και έχουμε, έχουμε φτάσει σε, στην τέταρτη φάση. Πρέπει εμεί να εξασφαλίσουμε να καλυφθούν οι ανάγκες τη αποστολή στο μέλλον. Πάντως, η συζήτηση ήταν ευρύτερη για ε, την αποστολή εκεί. Μας ενημέρωσε ο, ο Γάλλος υπουργό για τις συνεχείς προσπάθειές τους. Και από 4.000 που είναι η γαλλική δύναμη θα μειωθεί μετά το καλοκαίρι σε 2.000 και μετά τέλος του έτους θα ε, έχουν χίλιους άνδρες. Οπότε παράλληλα θα έχουμε και ανάπτυξη της αφίσμα που είναι η, η αφρικανική δύναμη και παράλληλα η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Αυτό από τον Ιούλιο. Βέβαια θα αναζητείται ακόμα η νομική βάση και υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή σήμερα κιόλα το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την νομική βάση και τα λοιπά μια που συνεχίζεται τώρα η συνεδρίαση στην Νέα Υόρκη συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ πάρα πολύ συχνά όσον αφορά το Μάλι για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ε, αυτή την, υποκατάσταση της μιας υποστολής από την άλλη να δούμε και οικονομικής πλευράς τι μπορεί να γίνει και γενικότερα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πέραν των οικονομικών. Οι υπουργοί επίσης ανέφεραν το τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και τις σχετικές υπηρεσίες. Κατά κάποιο τρόπο ε, μη στατιωτικού χαρακτήρα ε, προσωπικού ασφαλείας. Γιατί ξεκάθαρα η κυβέρνηση της χώρας μας είπε ότι προσδοκά να τους βοηθήσουμε όσον αφορά χωροφυλακή, αστυνομία, ε, αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οπότε και προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό και όλο αυτό αναφέρεται επίσης και στα συμπράσματα του Συμβουλίου της 22ης Απριλίου. Άρα θα έχει συνέχεια το θέμα και η πατεκπρόσωπος επίσης ενημέρωσε τους ε, Υπουργούς Αμήνης σε σχέση με τον διάλογο ε, Σερβίας Κοσόβου που είχε πάρα πολύ ευτυχή κατάληξη την Παρασκευή. Ε, γιατί αυτό θα έχει επιχειρησιακές συνέπειες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την, την ΚΕΙΦΟΡ και, το, και τις δυνάμεις του, του, του ΝΑΤΟ ε, που έχουν συμμετάσχει δια του αναπληρωτή ε, Γενικού Γραμματέα, του κ. Βέσπο, ο οποίος ήταν στο, στη συζήτηση αυτή που σας ανέφερα, το Συμβούλιο. Έχουμε τώρα το Συμβούλιο το οποίο διεξήφθησε δύο ημίση. Πρώτα-πρώτα συζητήθηκε το θέμα της υπηρεσίας ε, άμυνας και έχουμε τώρα τα νέα προγράμματα συνεργασίας ε, για την, ε, αντεονεφοδιασμό εφοδιασμό εν πτήση των αεροσκαφών. Επίσης συζητήθηκε η κυβερνό ασφάλεια, τα συστήματα που έχουν σχέση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και επίσης η προετοιμασία του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου όπου θα ζητούν τα θέματα αμήνης και ασφαλείας. Και θα επανέλθω σε αυτό. Ε, βέβαια στη διευθύνουσα ομάδα ξέρετε ότι υπάρχει ένα κατόπιν που δεν πηγαίνει. Κατόπιν είχαμε το σύνολο του Συμβουλίου όπου συμμετέσχουν όλα τα μέλη και εκεί έγινε μια μακροσκελή παρουσίαση από πλευρά του Επιτρόπου κ. Ταγιάννη όσον αφορά την Task Force για την άμυνα και την ε, προετοιμασία τη ε, ανακοίνωση τη Επιτροπή όσον αφορά την ε, αμυντική βιομηχανία και τα σχετικά με την αγορά. Από ό,τι ξέρω, σα ενημέρωσε χθε ο κ. Ταγιάννη. Πάντω, μα είπε πώ έχουν τα πράγματα, μα είπε τι δυνατότητε υπάρχουν όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία το ρόλο των ΜΜΕ και μας είπε ότι αναζητείται ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και των ιδιομορφιών ε, της βιομηχανίας αυτής και των σχετικών κρατικών προμηθειών. Βεβαίως και χρειάζεται όμως να υπάρχει μια στέρεη βάση για τη βιομηχανία μας στην Ευρώπη, εάν θέλουμε να εξελίξουμε τις ε, στρατιωτικές μας δυνατότητες με τρόπο βιώσιμο. Αυτό θα ωφελήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ. Άλλωστε μιλούμε για χώρες που συμμετέχουν και στους δύο φορείς. Επίσης κάποιοι υπουργοί ανέφεραν το θέμα της ε, εντολής για εμπόριο και επενδύσεις ε, και την υπερατλαντική μας εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Οπότε το θέμα είναι κατά πόσον η άμυνα θα καλύψει την εντολή. Είναι διχασμένα τα κρατημέλη σε σχέση με αυτό. Συνεχίζεται η συζήτηση. Απλώ σα επισημαίνω ότι πρόκειται κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλού. Και δεν θέλησε η πατικρόσωπο να το συζητήσει αυτό. Ε, αυτό είναι θέμα επίσης ε, των Υπουργών Εμπορίου. Απλώς αναφέρθηκε και σα το αναφέρω, γιατί προξένησε έντονο ενδιαφέρον. Επίσης, είχαμε μια σύντομη συζήτηση για τις ομάδες μάχης. Είπαμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει γιατί αυτό το θέμα εκκρεμεί εδώ και χρόνια, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτό το μέσο και είπαμε ότι θα πρέπει οι ομάδες μάχης να αποτελέσουν κομμάτι των επιχειρήσεων. Πολλά κράτη-μέλη τώρα έχουν επανέλθει με ιδέες για το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό το μέσο από Λιθουανία, Λετωνία, Ενωμένο Βασίλειο υπήρξαν προτάσεις και είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ε, ευέλικτη προσέγγιση και ε, από πλευρά επιμελητία, από πλευρά ιατρική κάλυψη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι ομάδε. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί πάντω η έννοια αυτή, ούτω ώστε η ομάδα μάχη να μπορέσει να παράσχει και κάποιε εκπαιδευτικέ δραστηριότητε στη Σομαλία, έχουν γίνει κάποιες αποστολές στο Μαλί και λέγεται ότι θα πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε. Ε, υπήρξε ανταπόκριση θετική και υπήρξε επίσης συζήτηση, είπαμε, στο Συμβούλιο, που θα ακολουθήσει τις αμέσως μέρες ή εβδομάδες. Να σας πω τώρα για κάθε αυτό το Συμβούλιο, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό θα είναι από πλευρά ΚΕΠΑ το γεγονός της χρονιάς, το πιο σπουδαίο. Το είπε και η, η εκπρόσωπος, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, χαρακτηριστικά. Οπότε είπαμε θα πρέπει να δούμε τι θα αποσπάσουμε από εκεί, όπως ας πούμε την ε, ανακοίνωση που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλές προτάσεις ε, θα κατεβάσει η Επιτροπή μέσω της ανακοίνωσης. Να δούμε επίσης πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως και Οπότε οπωσδήποτε είπαμε ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε καλύτερα τα χρήματα της ε, άμυνας. Και επίσης τονίστηκε ε, το τι θα γίνει με τις δυνατότητες μπορούμε να έχουμε ως και πά. Και από πλευράς τεχνολογίας ε, Σα έχει μιλήσει φαντάζομαι ο κύριος Σταγιάννη, όπως και συζητήθηκε, γιατί είπαμε εκεί υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για τη διπλή χρήση, πολλαπλή χρήση τέλο πάντων κάποιων προγραμμάτων. Ε, κυρίως όσον αφορά κάποια αεροσκάφη και άλλες συσκευές και είπαμε ότι μπορούν να έχουμε ερευνητικά προγράμματα ε, πολιτικού χαρακτήρα. Ας πούμε στα πλαίσια της πολιτικής ε, για το 2020. Αλλά και στρατιωτικού χαρακτήρα έρευνα. Προτυποποίηση, πιστοποίηση, πρόκειται για τομείς όπου μπορούμε να έχουμε μεγάλη οικονομία κλίμακος. Και αυτό επομένως θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάντως, αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε από τους ηγέτες αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων είναι ότι θα πρέπει να δώσουν μια κατεύθυνση μέσα των συζητήσεων για την μελλοντική ανάπτυξη της ΚΕΠΑ. Τι κατεύθυνση θέλουν να πάρει. Πώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε τον ρόλο μας ως πηγή και πάροχη ούτως υπήν ασφάλειας. Κάποια κρατημέλη είπαν ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε την υπάρχουσα. Υπάρχει εκεί πέρα κάποια διχογνωμία, άρα και δεν καταλήξαμε πουθενά. Επομένω δεν έγινε συζήτηση κατέληξε κάπου. Πάντω χρειάζεται να υπάρχει στρατηγικό προσανατολισμό υψηλού επίπεδου. Πάντω η ζήτηση δεν θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. θα χρειαστεί να γίνει σύνθεση βέβαια για να πάμε κάπου και επομένω θα υπάρξουν κάποια πρακτικά διαβήματα ε, όπως είπε και ο Επίτροπος Ταγιάννη θα έχουμε τέλη Ιουνίου την έκθεση της ε, εκπροσώπων εκπροσώπου όσον αφορά ε, Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο τέλο πάντων θα, θα γίνει αυτό όσον αφορά τις θέσεις της υπάντης εκπροσώπου για το Συμβούλιο, επί τη βάση των το τελευταίο Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο και ο πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Φανεροπάη θα διατυπώσει τι δικέ του συστάσεις και και κάποιο σχέδιο συμπερασμάτων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Οπότε έχουμε τώρα τι διάφορε ομάδε θεμάτων που θα ζητηθούν από υψηλούς αξιωματούχου, από του υπουργού Άμυνα. Ε, από τώρα μέχρι και τότε το τέλος του έτους. Thank you. My colleague. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλουν συνάδελφοι να υποβάλουν ερωτήσεις. Ορίστε. Έχ... Κυρία Γκουράκη, έχετε το λόγο. Ε, ε, ε, έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το τελευταίο κομμάτι που μας είπε ε, μας είπατε και αφορά την, ε, τη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο για την ΚΕΠΑ. Ε, είπατε ότι υπήρχαν... Ε, there is no translation. Yeah, kind Okay. Uh, so I, I'm starting again. So I, I have some questions. Έχω μερικές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη συζήτηση που έγινε στην ΚΕΠΑ, στη, στο Συμβούλιο για την κατεύθυνση της ΚΕΠΑ. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι υπήρχαν κάποια, κάποιες χώρες μέλη που θέλανε μία αλλαγή στη στρατηγική. Μήπως μπορείτε να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένος ε, στο ζήτημα αυτό. Έχει αυτό να κάνει με αυτό που είδα στην ομιλία του, του Προέδρου, του κυρίου Ρομπάη, ότι θεωρεί στην άμυνα ότι υπάρχουν δύο καινούργια στοιχεία ότι η άμυνα πλέον δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς και η άμυνα είναι άειλη, δηλαδή μια, μια αντίληψη που για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με τα battle groups. Έγινε καμιά συζήτηση για μείωση του ορίου επέμβασης αυτών των δυνάμεων. Γιατί ως γνωστόν υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν χώρες που θέλουν πιο γρήγορα να επεμβαίνουν τα battle groups, κάποιες ε, όχι και υπάρχει ένα όριο. Έγινε κάποια συζήτηση στο ζήτημα αυτό. Τρίτο ζήτημα ε, για τη Συρία. Δεν υπάρχει τίποτα στο κοινό ανακοινωθέν, στα, συμπεράσματα, όμως ε, παίρνω την ε, τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος κάτι είπε για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι, έγινε καμιά συζήτηση για αποστολή εξοπλισμού ή άλλου είδους υλικού ε, στους ε, ε, αντιφρονούντες στη Συρία. Υπήρχε κάτι πέραν αυτών που διαβάσαμε για το πετρέλαιο και για τους πρόσφυγες στη Ιορδανία και στη, στο Λίβανο. Εμένα με ενδιαφέρει στο εξοπλιστικό. για το Κόσοβο είχα διαβάσει ότι η, η Σερβία ε, δεν θα δεχτεί ε, το Κόσοβο να είναι στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά. Μετά τις συνομιλίες μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, που συμφωνήσαν σε αυτά που συμφωνήσαν, ε, εκ μέρους της σερβικής πλευράς υπόθηκε ότι η Σερβία δεν θα αναγνωρίσει το Κόσοβο σε διεθνείς οργανισμούς. Ξέρετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε. Και αν τελευταία αφορά το Μάλι, και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την υπομονή σας στο σημείο 12 του ανακοινωθέντος για το Μάλι στο σημείο 12 ε, γίνεται λόγος για κάποια μέτρα γίνεται λόγος για μέτρα στις χώρες που συνορεύουν με το Μάλι για μέτρα ασφάλειας ως ε, συνέπεια των κινδύνων που, έχουν δημιουργηθεί, που έχει δημιουργήσει η κατάσταση στο Μάλι. Δηλαδή στο σημείο 12 των συμπερασμάτων για το Μάλι γίνεται λόγος για συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν απειλές σε γειτονικέ χώρες του Μάλι που δημιουργήθηκαν από την κατάσταση στο Μάλι. Περί τίνος πρόκειται, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις και ίσως ερωτήσεις. Βλέποντας λοιπόν το πρόγραμμα των συζητήσεων για την ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι έχουμε τεράστια προβλήματα. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε τις προτεραιότητες που τίθενται για την πολιτική μας. Λιβύη. Η μελλοντική αποστολή για την εκπαίδευση της ακτοφυλακής. Πριν από μερικές εβδομάδες. Στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε τον πρώην ηγέτη του Προσωρινού Συμβουλίου, τον κύριο Τζαμπρίλ. Έθεσε το πρόβλημα. Τεράστιος όγκος όπλων παραμένει στα χέρια του πληθυσμού της Λιβύης. Το θεωρούν προτεραιότητα το ζήτημα. Διότι αυτά τα όπλα οδηγούν, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικά δίκτυα επίσης. Όχι μόνο τη σταθεροποίηση της χώρας. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Σαχάρα και στο Μαλί. Εντοπίζουμε σαν προτεραιότητα ε, για τη Λιβύη τα σύνορα. Και έχουμε και στην ενδοχώρα τεράστια προβλήματα. Τώρα τα battle groups δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ αυτές οι μονάδες, οι μάχοι Προσπαθήσαμε να μοιραστούμε το κόστος προετοιμασίας, εκπαίδευσης και ασκήσεων, αλλά δεν βλέπω συγκεκριμένη απόφαση. Και πώς θα εφαρμοστεί, θα λειτουργήσουν αυτά τα battle groups. Είναι κρίσιμα για την ε, ΚΕΠΑ, πιστεύω εγώ. Τίποτα άλλο όμως δεν έχει προσθεθεί σε αυτά που ξέρουμε. Γιατί έχουμε τις μονάδες. Τα χρειαζόμαστε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μονάδες τελικά, τις battle groups. Μετά το Μάλι ξεκίνησε μια αποστολή Ο επικεφαλής ήδη αναφέρθηκε την επόμενη φοιτεία. Δεν εγκρίνει τον τρόπο εκπαίδευσης. Γίνεται προσπάθεια ανοικοδόμησης του στρατού του Μάλι Αλλά όχι η υποστήριξη αποστολών ή προστασία αποστολών, αλλά για την ανοικοδόμηση και την αδιάθεση του στρατού. Εκεί δίνεται προτεραιότητα. Αυτό μα δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τι προτεραιότητε τη ΚΕΠΑ. Και υπονομεύει αυτό ο κίνδυνο κάπω την. Αυτή η έλλειψη προτεραιοτήτων υπονομεύει τελικά την επίτευξη των στόχων τη ΚΕΠΑ. Η κυρία Γκόμε, δεν θέλω να ξεκινήσω συζήτηση τώρα, δεν υπάρχει χρόνος. Κύριε Ποπόσκι, για την επόμενη φορά θέλω να θέσω κάποια πράγματα. Ήρθα από τη Λιβύη, το Σαββατοκύριακο μου στη Λιβύη, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Σύντομα θα στείλω άτυπη έκθεση που αφορά την έκθεση. Όλοι οι συνομιλητές μου στη Λιβύη και Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Δικαιοσύνη, αλλά και βουλευτέ, μου τόνισαν τη σημασία που προσδίδουν στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συλλογή των όπλων και την δόμηση δομών ασφαλείας, αστυνομίας δηλαδή και στρατού πέρα από την προστασία των συνόρων. Ξέρω ότι η ασφάλεια των συνόρων που προσφέρεται και υποστήριζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που χρονολογείται πίσω στη διάσκεψη εκεί που ανετέθη αυτό στα πλαίσια των συζητήσεων. Πρέπει να εφαρμόσει την ασφάλεια των συνόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποστολή αρχίζει και οργανώνεται εκεί. Για το θέμα της ασφαλείας των συνόρων ε, υπάρχουν πέντε άνθρωποι εκεί. Τον Ιούνιο θα λειτουργήσει το σύστημα. Μου είπαν ότι πιθανότατα δεν θα λειτουργήσουν όλα σωστά ε, πριν τον Νοέμβριο. Είναι η αποστολή της ΚΕΠΑ που αφορά την προστασία των συνόρων. Τι συμβαίνει στη Λιβύη. Δεν αφορά τη δική τους ασφάλεια των Λιβύων, αλλά τη δική μας ασφάλεια. Τα είδαμε με την απόπειρα, την επίθεση κατά της γαλλικής πρεσβείας. Το ότι αυτές οι πολιτοφυλακές είναι ο μόνος μηχανισμός ασφαλείας και δέχονται δίσδυση από τους τζιχαντιστές που στηρίζονται με τα χρήματα. Μπορούμε να μαζεύουμε τα όπλα, αλλά μπορούν να βρουν καινούργια όπλα. Γιατί παντού στη Λιβύη υπάρχουν όπλα. Που έρχονται απ' έξω, κυρίως από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο πολιτικό και βέβαια και όσον αφορά την ασφάλεια. Και γι' αυτό όλοι στη Λιβύη, όλος ο κόσμος μας ρωτάει, μας ζητά, κάντε κάτι. Γιατί εμείς διστάζουμε. Γιατί η Λέβη Άστον δεν αναλαμβάνει να πείσει τα κράτη-μέλη μας να κάνουν μια κανονική αποστολή ΚΕΠΑ στη Λιβύη που προχωρά πέρα από την φύλαξη των συνόρων. Κάτι που πρέπει να οργανωθεί με τις λιβικές αρχές. Αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Μας το ζητούν. Αυτό αφορά την ασφάλειά μας. Ευχαριστώ, Άννα. Ήρθε η ώρα για απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις. Για το πού πηγαίνει η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τι θέλουν να αλλάξουν οι χώρες μέλη. Ίσως ακούσατε από τον Καρλ Μπίλτ, που είναι μεγάλος υποστηρικτής μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής ε, ασφάλειας και αμυνάς. Νομίζω μίλησε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Για πολλούς απλώς σημαίνει μια επικαιροποίηση, διότι η αρχική ε, έγινε το 2003, επομένως είχε συνταχθεί σε μια άλλη εποχή η βασική της ανάλυση στην οποία στηρίζεται δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει βέβαια κατά τη γνώμη μου. Άλλες χώρες μέλη δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό αυτό και γνωρίζουν ότι η σύνταξη μιας νέας στρατηγικής ασφάλειας και άμυνας θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και κοπιαστική και μπορεί και να μην καταλήξει και πουθενά. Γιατί ποικίλουν και οι αντιλήψεις περί Απειλή και κινδύνου. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι κάποιο προβληματισμό για το πού θέλουμε να πάμε με την ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνα ω πολιτική, αντί να περάσουμε από μια διαδικασία σύνταξη νέου εγγράφου. Ο Καλ και επιτρέψτε μου να παραθέσω αυτό που είπε, γιατί το πιάσε σωστά, είπε η διαδικασία έχει περισσότερη σημασία από την έκβαση. Συμφωνώ μαζί του. Ο πρόεδρος Βαν Ρόμποϊ, μάλλον αναφέρεστε στην ομιλία του στην ε, ετήσια διάσκεψη της κοινότητας ασφάλειας και άμυνας, αλλά μίλησε με ευρία έννοια. Αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον ίδιο είναι η κατάσταση της άμυνας στην Ευρώπη και όχι μόνο η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αναφερόταν δηλαδή και στην κατάσταση της ευρωπαϊκής ε, αμυντικής βιομηχανίας, Τη αμυντική, τη αγορά άμυνας δηλαδή, και επίσης όπου η αμυντική βιομηχανία έχει και άλλες πτυχές που είναι πολύ σημαντικέ για τους Ευρωπαίους ηγέτε. δηλαδή ανταγωνιστικότητα, δημιουργία απασχόλησης, δημιουργία αξίας στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να προσεγγίσει τη συζήτηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα, όρια για τις παρεμβάσεις των ε, μάχημων ομάδων. Υπάρχουν πρώτα-πρώτα οικονομικά όρια. Είναι δηλαδή ένα είδος αντικίνητρα για τις χώρες μέλη το υψηλό κόστος. Για τις χώρες δηλαδή που διαθέτουν δυνάμεις στις ε, μάχημες ομάδες. Είναι βέβαια και πρωτίστως θέμα πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει οι χώρες μέλη να έχουν την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσουν τις ε, battle groups, τις οι battle groups ως έννοια ξεπήδησαν μέσα από μια πρακτική εμπειρία. Την πρώτη ευρωπαϊκή επιχείρηση σε αφρικανικό έδαφος στη Δημοκρατία του Κονγκό το 2003. Δεν ήταν μάχημη ομάδα τότε, αλλά την εμπειρία εκείνη θελήσαμε να τη βάλουμε σε ένα κόνσεπτ, σε μια αντίληψη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Αλλά όπως είπα πριν, έχει έρθει η ώρα να πάρουμε απόφαση εάν όντω θέλουμε να τις χρησιμοποιούμε με επιχειρησιακό τρόπο ή όχι διότι έχει ήδη κάποια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, καλύτερη διαλειτουργικότητα, επίσης βελτίωση της εκπαίδευσης των ε, δυνάμεων. Αλλά επιχειρησιακά δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Ούτε έχει γίνει καμιά ειδική συζήτηση μεταξύ Υπουργών Άμυνας για τη Συρία. Ακόμα συζητιέται ε, στους Υπουργούς Εξωτερικών, οι οποίοι θα επανέλθουν στη διάσκεψη του Μαΐου και το εμπάργο όπλων λύγει τον Ιούνιο. Οπότε θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουν και να λάβουν νέα απόφαση. Και όπως σωστά είπατε, λήφθηκε η απόφαση να επιτραπεί η αγορά πετρελαίου από τις πηγές που, ελέγχει, που ελέγχουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η μόνη πτυχή που συζητήθηκε. Τώρα, Σερβία Κόσοβο δεν συζητήθηκε, προσπαθώντας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της συμφωνίας μεταξύ Σερβίας Κωσόβου της προηγούμενης Παρασκευής, όπου και οι δύο πλευρές είπαν δεν θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ανέλαβαν τη δέσμευση να μην κάνουν οτιδήποτε, να μην πράξουν τίποτε που θα υπονομεύσει την διαδικασία ένταξης της άλλης μεριάς αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση για άλλο διεθνή οργανισμό. Δεν μπορώ λοιπόν να σχολιάσω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Τώρα για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Μάλι και μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν για ή σε γειτονικέ χώρε. Αυτό συνεχίζεται εν μέρη με εμπλοκή στη Λιβύη. Θα απαντήσω όμως μετά γι' αυτό στην κυρία Γκόμες. Βέβαια πρέπει να εξετάσει κανείς την περιοχή αυτή ως σύνολο. Ήδη βρισκόμαστε στον Νίγηρα. Έχουμε αρχίσει δηλαδή εκπαίδευση εκεί των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων της χωροφυλακής στον Ήγηρα πριν από λίγους μήνες. Αυτό κάπως επισκιάστηκε από την εξέλιξη στο Μάλι, αλλά υπάρχει δουλειά που γίνεται εκεί από ανθρώπους επιτόπου. Η δε εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης για το Σαχέλ προβλέπει και άλλα μέτρα, κυρίως μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά συζητούμε τώρα με την Κομισιόν για τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης για τα 7 χρόνια μετά το 2014 και ορισμένες από τις χώρες αυτές θα γίνουν και κύριοι τομείς ε, για την ασφάλεια στη Σαχέλ. Αν μπορώ τώρα να συνδυάσω και με τα σχόλια της κ. Νικολάη για τη Λιβύη. Το θέμα των όπλων είναι πραγματικό. Κάποια στιγμή στο παρελθόν χρησιμοποίησαμε κάποια από τα μέσα που έχουμε στον προπολογισμό μας για σταθερότητα για να προβλέψουμε καλύτερη φύλαξη στις αποθήκες όπλων. αλλά δεν είναι πλήρης βέβαια η φύλαξη αυτή και χρειάζεται να το ξαναδούμε. Η εμπλοκή περιορίζεται για την ώρα στην ε, αποστολή συνόρων. Δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί η αποστολή αυτή. Γνωρίζετε και το ιστορικό, πόσο χρειάστηκε, πόσα, πόσο χρόνο χρειάστηκε. Διαπιστώσαμε πάλι ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στους κανονισμούς μας που καθυστέρησαν την ανάπτυξη της αποστολής, αλλά υπάρχει όταν και έφτασε στην Τρίπολη την προηγούμενη εβδομάδα και ε, λαμβάνει ενεργό ε, μέρος στο σχεδιασμό και θα ολοκληρωθεί μέσα με τέλη Ιουνίου και μετά θα αρχίσει να εργάζεται. Οι συνθήκες ασφαλείας ωστόσο είναι αυτές που είναι. Γνωρίζουμε τι έγινε την Δευτέρα. Σοβαρότατη επίθεση κατά της γαλλικής πρεσβείας και λαμβάνουμε εκεί υπόψη βέβαια και τις επιπτώσεις στο δικό μας το προσωπικό. Μόλις έλαβα μήνυμα από τον αναπληρωτή μας επικεφαλής αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με όλους τους Ευρωπαίους πρεσβευτές σήμερα, μάλιστα αργότερα σήμερα, για να συζητήσει τις ε, περιστάσεις. Γιατί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή την ομάδα μας στη διαχείριση των συνόρων σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή κίνδυνη. Δεν το αποκλείουμε να αναπτυχθεί, αλλά για την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε στο core business, δηλαδή στα, στα απόλυτα απαραίτητα σημεία της αποστολής μας. Δεν έχει διεξαχθεί καμιά συζήτηση για χρήση των battle groups στο πλαίσιο αυτό. Ούτε θα είχε καμιά μεγάλη χρησιμότητα να χρησιμοποιηθούν οι battle groups ή τμήματά τους στη TV, γιατί δεν είναι κατάσταση μάχης. Χρειάζεται να γίνουν κάποια σταθεροποιητικά και χρειάζεται και πραγματική αναδιάρθρωση του τομέα της ασφάλειας. Πρέπει ταυτόχρονα ωστόσο να σχεδιάσουμε για πολλά ενδεχόμενα. Επίσης έχουμε ενισχύσει την ομάδα μας επιτόπου, την αντιπροσωπεία δηλαδή, με εμπειρογνώμονες ασφάλειας, αστυνομίας και χωροφυλακής. Βρίσκονται εκεί ως σύμβουλοι της ομάδας μας και συνεργάζονται με τους διάφορους, ε, με διάφορους οργανισμούς στη Λιβύη. Η κυβέρνηση για την ώρα είναι σταθεροποιημένη, γιατί ήταν και δύσκολο να βρούμε συνομιλητές. Ε, Πριν 1,5 χρόνο είχα βρεθεί ο ίδιος εκεί και ε, έκανα πολύ χρήσιμες συζητήσεις με ορισμένα στελέχη, λιβικά στελέχη δηλαδή, που μετά από δύο εβδομάδες είχαν φύγει από τις θέσεις τους. Είχαν παθεί για το Μάλι. Δεν συζητούμε για την επόμενη ε, εντολή. Η εντολή μας διαρκεί 15 μήνες. Δεν νομίζω ότι θα αρκέσουν, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτά πρέπει να κάνουμε. Αλλά η εντολή είναι πολύ σχηδής. Όχι μόνο για την βασική στρατιωτική εκπαίδευση των δυνάμεων του Μάλι, τέσσερα τάγματα έχουν, αλλά και παροχή στρατηγικών συμβουλών στις ένοπλες δυνάμεις, του Μάλι και την αναδιάθρωση του στρατού τους. Γνωρίζω ότι έγιναν και κάποια σχόλια στον τύπο για την κατάσταση του στρατού του Μάλι. Πράγματι έχει υποστεί πολλά δυνά ο στρατός αυτός. Θα πρέπει να ξαναβρεθεί σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι ένας από τους κύριους στόχους της εκπαιδευτικής μας αποστολής επιτόπου. Και ένα σημαντικό καθήκον είναι και η παρακολούθηση βέβαια της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της τήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Μάλι από όλες τις πλευρές της σύγκρουσης. Έχουμε λοιπόν αυτό τον ορίζοντα των 15 μηνών και πρέπει ασφαλώς να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Θα γίνει μια έκθεση στους έξι μήνες, κάποια στιγμή το φθινόπωρο, και είμαι βέβαιος ότι οι Υπουργοί Άμυνας θα επανέλθουν να επανεξετάσουν τη συζήτηση στην επόμενη, στο επόμενο Συμβούλιο τους, νομίζω τον Νοέμβριο φέτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώσαμε το θέμα σήμερα. Επόμενη συνεδρία στις 16 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Μάλι θα είναι εδώ και η δεύτερη συνεδρίαση 20 Μαΐου στο Στρασβούργο με το Γάλλο Υπουργό Άμυνας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Γεια σας.